Σε όλο αυτό το πελώριο έργο προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία φυσικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε. Ε, συνάδελφοι, λίγη η συζήτηση για αυτό το θέμα. Αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Και τώρα... Περνούμε στην τελευταία έκθεση της ε, σημερινής ε, συνόδου, η έκθεση της κυρίας Μαρία Νταγκράσα Καρβάλιο, εφαρμογή των προγραμμάτων πλαίσιο έρευνας. Η συγγήτριά μας ε, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η επιστήμη, η καινοτομία και η τεχνολογία είναι οι βασικοί πυλώνες της ε, ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο, να ανοίξει τα συστήματα έρευνάς της να βοηθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, επιστημόνων και να προωθήσει την αριστεία. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι όλο και πιο πολυπολικός και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την επιστήμη. Αρκεί να αναφέρω ορισμένου αριθμού, ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. 80% των επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο εργάζονται έξω από την Ευρώπη και 79% των ευρεσιτεχνιών καταγράφονται εκτός Ευρώπη η Ευρώπη δε υπολείπεται της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε επένδυση και αυτό κυρίως οφείλεται στην έλλειψη επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τα συστήματα καινοτομία και επιστήμης, να ξεπεράσουμε την υποχρηματοδότηση, τον κατακαιρματισμό, την έλλειψη δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την καινοτομία και την υπερβολική φυσικά γεωγραφία. Το ευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να ξεκινήσουμε την απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης για να μεταρρυθμιστεί. Και γι' αυτό εγώ ως εισηγήτρια θέλω να ζητήσω να απλοποιηθούν οι κανόνες για τη συμμετοχή σε τωρινά και μελλοντικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας. Η έκθεσή μου θέλει να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί βρισκόμαστε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του 7ου προγράμματος πλαίσιου για την έρευνα και την ανάπτυξη και της προετοιμασίας του 8ου τέτοιου προγράμματος. Εγώ ως εισηγήτρια στέλωσα να ξεκινήσω μια συζήτηση για τα θέματα αυτά και να κάνω μια δημόσια διαβούλευση να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή όλων των φορέων. Υπήρξε πράγματι σε αυτή τη διαβούλευση ένας μεγάλος αριθμός συμβολών που κατέληξε ότι οι πολίτες μας και τα κράτη μας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την έρευνα. Τονίζεται η ανάγκη να απλοποιηθούν οι ελεκτικές διαδικασίες και να υπάρξει μια πιο απλή διαδικασία Αξιολόγηση από τους ομοτήμους επί τη βάση της αριστείας. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή στον κίνδυνο, να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί ελέγχου και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην επιστημονική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά η έκθεση αυτή είναι απλώ η απαρχή μια διαδικασία η οποία δεν θα είναι απλή. Η εφαρμογή αυτών των συστάσεων θα πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι απαραίτητο να υπάρξει πολιτική υποστήριξη και παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να μπορέσει να έρθει σε αίσιο πέρας και ασφαλή λιμένα αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία της απλοποίησης θα πρέπει στο μέλλον να επεκταθεί και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδίως στα διαρθωτικά ταμεία. <clears throat> προγράμματα με απλούστερους κανόνες και θα είναι συγχρόνω και πιο αποτελεσματικά και πιο διάφανα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλου τους συναδέλφους μου και τη Βελγική Προεδρία, την Κομισιόν, ε, και όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν, χώρα, έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση. Το να απλοποιήσουμε σήμερα την πρόσβαση στα δημόσια κονδύλια για την ε, επιστήμη και την ανάπτυξη, αυτό θα οδηγήσει σε μια εταιρική σχέση στο μέλλον από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων και με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η έρευνα και η καινοτομία στην Ευρώπη και έτσι η Ευρώπη θα γίνει ένας ελκυστικός χώρος για να ζει κανείς, να εργάζεται και να είναι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Θα αρχίσει η οφθαλμοθυρία. Η κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας για τη δουλειά που έκανε, διότι η απλούστευση της εκτέλεσης των προγραμμάτων πλαίσιο για την έρευνα είναι μια αναγκαιότητα. Και όπως είπε σωστά η συγγήτριά μας, αυτό είναι μόνο μία από τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και ε, πιο πολυσχηδής ε, και να τονώσει την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Ε, κρατάει η συγγήτρια το αρχικό πεδίο εφαρμογή τη προ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνούμε και έχει προτάσει για τη χρηματοδότηση, για την απλούστευση του μέσου κόστου εργασία, το μηχανισμό καταγραφή των ωραρίων, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να επιμείνουμε για την ε, επιστροφή των εξόδων των συμμετεχόντων, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, ακαδημαϊκών, γιατί αυτοί είναι οι πυλώνες της ε, ανάπτυξης ε, και της οικονομικής ευημερίας. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε τις προτάσεις της έκθεσης και να προαγάγουμε έτσι την έρευνα και την επιστήμη. Mm. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία. Εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαβιβάστε και τις ευχαριστίες μου στην κυρία Γκέγαν Κουίν ε, γιατί προώθησε τα περί και κωδικοποίησης. Πρέπει να απλουστεύσουμε το μέλλον μας. Αλλά πρέπει να κλείσουμε και τους παρελθόντους λογαριασμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ναι, πρέπει να εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες από αυτού που είχαν εγκριθεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν πριν προχωρήσουμε. Έχουμε φτιάξει ερευνητικά Ινστιτούτα που δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα ε, ε, τηρώντας ε, την χρηστή διαχείριση και με τα ανεκτά ποσοστά λάθους αλλά και χρησιμοποιώντας εξωτερική πραγματογνωμοσύνη και ενδεχομένω, όπως πρότεινα και έγινε δεκτό με έναν ανεξάρτητο μερόληπτο διαμεσολαβητή πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ερευνητικών Ινστιτούτων με καλούς ελέγχους βεβαίως με χρηματοδότηση της Ένωσης έτσι θα εισέλθουμε στις διαπραγματεύσεις των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών ούτως ώστε να ε, ε, καταστήσουμε πιο ε, ευρωπαϊκή την έρευνα στην υπηρεσία φυσικά των πολιτών της Ένωσης. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρίσα Ματίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Γκράσσα Καρβάλιου για τη θαυμασία έκθεση που μας παρουσίασε και να τονίσω ότι η διαδικασία αυτή έγινε πραγματικά με πολύ δημοκρατικό τρόπο και εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό και πάλι εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Έχουμε ένα από τα πιο ευραία προγράμματα έρευνα και ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα έρευνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρόταση τη κυρία Καρβάλιου εμπλουτίζει ιδιαίτερα την πρόταση τη Κομισιόν κατανοεί ότι δεν αρκεί μονάχα η απλοποίηση, ότι είναι σημαντική η αξιολόγηση όλων των φορέων ε, της ε, ανάπτυξης, προωθεί τη συμμετοχή, τη δημοκρατία και τη διαφάνεια μέσα σε ένα πλαίσιο ισότητας ευκαιριών, ευκαιριών για όλους. Να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο δεν βασίζεται στο γραφειοκρατικό έλεγχο, αλλά βασίζεται στην ανεξαρτησία της ε, έρευνας και την αναγνώριση της συνεργασίας διαφόρων επιστημονικών τομέων και της αξιολόγησης από ομότιμους. Για όλους αυτούς τους λόγους και κλείνω κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η εφαρμογή αυτής της πρότασης κυρίας Καρβάλιο θα βελτιώσει τα μάλα της συνθήκες εργασίας όλων των ερευνητών στην Ευρώπη και θα, άρει, θα εξάρει το ρόλο τους και θα αυξήσει την αξιοπρέπεια τους και πρέπει όλοι από κοινού να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ε, Πολύ εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τον υπερβολικό ανταγωνισμό που υπάρχει. Παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων δεν υπάρχει πλήρης πρόσβαση για όλους παρά την εργασία που μπορεί να έχουν επιδείξει για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους του 2020 για τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% ε, θα πρέπει εγώ νομίζω να το κάνουμε 50% αυτό γιατί από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει μια αίτηση μέχρι να εγκριθεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει αυτοκαταργηθεί αυτό λόγω των δυσκολιών που του τίθενται λόγω της πολυπλοκότητας των μηχανισμών. Χρειάζεται οπωσδήποτε απλοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη. Κυρία Επίτη εσείς θα μας τελειώσετε τη συνοδό μας. Θέλω να σας συγχαρώ και εγώ κυρία Καρβάλιο για αυτή την έκθεση και για μας τίθεται το θέμα ιδίως στον τομέα της έρευνας, της πολυπλοκότητας και άρα της απλοποίησης. Έχουμε κάνει μία σχετική ανακοίνωση φέτος όπως γνωρίζετε με πολλές εναλλακτικές λύσεις για απλοποίηση, πράγμα το οποίο οδήγησε σε μια διαθεσμική συζήτηση για την οποία είμαστε ευγνώμονες και προς το Κοινοβούλιο. Καθώς και για την έκθεσή σας βέβαια που υποστηρίζει τις περισσότερες από τις προτάσεις μας, αν και οι δικές σας δεν είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες. Το Συμβούλιο ελπίζουμε να εγκρίνει και αυτό την ευρεία αυτή η συνένεση και να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε στην πράξη. Είμαστε υπέρ της απλοποίησης και των αρχών, που αναφέρεται, των αρχών της που αναφέρεται στην έκθεσή σας διαφάνεια, νομική σαφήνεια, βεβαιότητα και μία προσέγγιση που να βασίζεται περισσότερο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μερικές από τις προτάσεις σας όπως και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στο υπάρχον πλαίσιο αλλά εμείς ζητούμε και λύσεις που να μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα χωρίς υπερβολικό κόστος και χωρίς να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν εφαρμόσαμε το, πρόγραμμα, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, είχαμε ζητήσει να υπάρξει μια πιο ομοιογενής και συνεπής εφαρμογή των κανόνων, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ της υποβολής μιας αίτησης μέχρι τη χορήγηση του ποσού ή την εφαρμογή του προγράμματος. Και ξέρουμε ότι μόνο αν υπάρχει πραγματική απλοποίηση θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε ορισμένους από τους φραγμούς που τίθενται στην έρευνα. Έχουμε προβλέψει μηχανισμούς για τη διόρθωση λαθών ώστε να περιοριστούν αυτά σε κάτω από το 2%. αυτά που λέτε και εσείς για την διόρθωση των λαθών χωρίς υπερβολικό κόστος είναι πράγματα που τα δεχόμαστε. Με βάση βέβαια αυτή την περισσότερη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ερευνητών και ερευνητριών. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη σημαντικότατη αυτή σας έκθεση. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. και αυτή η συζήτηση θα ψηφίσουμε αύριο. Αύριο στις 9 θα ξαναρχίσει η σύνοδος, η Ολομέλεια και τα πρακτικά θα τα βρείτε στις ιστοσελίδες κλπ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας, ευχαριστώ και τις διερμηνές.